Οπότε θεωρούνται ως συγκεκριμένα τα πρακτικά. Και περνάμε στην έκθεση του κυρίου Σαλαφράγκα για τον ειδικό εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριε Σαλαφράγκα, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πατή Εκπρόσωπε, Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Παρά τη χρηματοπιστωτική κρίση, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το σχέδιο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης στηρίζεται σε αξίες, την ειρήνη, την κατανόηση, την ομόνια, την συμφιλίωση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που είναι εγγεγραμμένα στο γονιδίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στο γονιδίωμα και στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στο διατακτικό της συνθήκης της Λισαβόνας και στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εντός των θεσμικών οργάνων φυσικά ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό που κατεξοχήν έχει δεσμευτεί υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και έχει μία δέσμευση ακλόνητη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δεν θα πρέπει να αποτελούν προνόμιο μόνο μια περιοχή ή μια υπήρου, αλλά θα πρέπει να έχουν έναν οικουμενικό, διαπλανητικό χαρακτήρα. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέθεσε σε έναν αντιπρόεδρο το θέμα της, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα πλαίσια της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχουμε στήσει μια νέα ομάδα εργασίας για τη δημοκρατία και την παρακολούθηση των εκλογών. Και πάντα στις ημερήσεις διατάξεις μας έχουμε ηθικό κεφάλαιο για ε, θέματα προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχετικά ψηφίσματα. Και μάλιστα διακριθήκαμε με την απονομή βραβείου Ζαχάροφ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένα βραβείο για την ελευθερία συνείδησης που έχει ιδρυθεί από κάποιον που άφησε ένα σημαντικό κληροδότημα υπέρ της ειρήνης, του σεβασμού, της ανοχής και της αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ των λαών. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν κυρία Πρόεδρε χαίρομαι γιατί Υποβάλλω αυτή την έκθεση που με τη μορφή της σύστασης προς το Συμβούλιο αναφέρεται στο διορισμό του ειδικού εκπροσώπου ή εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της ε, πολιτικής μου ομάδας αλλά και τους συναδέλφους στην Επιτροπή Εξωτερικών. Ένα σημαντικό θέμα, κυρία είπατε εκπρόσωπε, είναι το θέμα της εντολής αυτού του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση και τη σφυριλάτηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, της ε, διεθνούς δικαιοσύνης και του ανθρωπιστικού δικαίου, υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής, να ασχοληθεί με δραστηριότητε για την προάσπιση των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, να καταπολεμήσει τα βασανιστήρια και την ατιμορρησία, να προαγάγει τα δικαιώματα των γυναικών, των μειονοτήτων, των παιδιών και την ειρήνη, την ασφάλεια και φυσικά να απορρίψει οποιαδήποτε μορφή διακριτική μεταχείριση. Αυτό ο ειδικό εντεταλμένο Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να συνεργάζεται άμεσα και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με άλλους διεθνείς οργανισμούς και να εξασφαλίσει σημαντική προβολή, ε, ελαστικότητα αλλά και συνέχεια με τις προηγούμενες μας δραστηριότητες. Θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να έχει πλούσια πείρα, προσόντα, ικανότητες, διεθνές κύρος και έγκλη και φυσικά γνώσεις στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σημαντικές επιδόσεις στον τομέα αυτό. Είναι ε, σημαντικό ότι δεν θέλουμε ε, να σφετεριστούμε τις ε, εξουσίες για τη λήψη αυτής της απόφασης, γιατί αρμόδια αυτό είναι η πατή για και το Συμβούλιο. Θα ήθελα όμως να τονίσω από την άποψη αυτή την ιδιαίτερη σημασία που έχει ο διορισμός αυτού του ειδικού εντεταλμένου και να εκφράσω επίσης την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση την εμπιστοσύνη και την εντολή που θα δώσουμε με το ψήφισμά μας ε, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο διορισμό αυτού του ανθρώπου που θα έχει τεράστια προβολή σε ό,τι αφορά την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα θέμα ιδιαίτερα προσφυλέ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μια σημαντική ακλόνητη δέσμευσή μα υπέρ των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Ευχαριστώ. Είπατε εκπρόσωπο. παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον κύριο Σαλανφράγκα ότι αυτό το θέμα είναι γεγραμμένο στο γονιδίωμά μα. Και μεγάλη χαρά χαίρομαι που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω στο Κοινοβούλιο για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπω ξέρουν οι βουλευτέ, είναι μία από τι ύψιστε προτεραιότητέ μου αυτή και κάθε ευκαιρία τη χρησιμοποιώ για να συνεχίσουμε τι συζητήσει μα. Ευχαριστώ λοιπόν επίσημα, κύριε Σαλαφράγκα, για τη δουλειά που κάναμε και κάνατε από αυτή τη έκθεση. Η σύσταση που έχετε ενώπιό σα είναι μια συνεισφορά στι προετοιμασίε για τον διορισμό ενό ειδικού εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είναι ο υπερασπιστής αυτής της ιδέας ε, με την έκθεση που συνέταξε το 2010. Φτάσαμε τώρα σε μια χρονική στιγμή όπου υπάρχει ευρεία συνένεση ε, σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Σας συγχαίρω κύριε Σαλαφράγκα που πετύχατε ε, μια τόσο, ένα τόσο καλό αποτέλεσμα της προφορίας στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Είναι αποτέλεσμα μιας ευρείας διαβούλευσης τους τελευταίους μήνες. Ήρθατε σε επαφή με, με μένα, με τις ε, υπηρεσίες μου, με τις υπηρεσίες της Κομισιόν και με, ε, με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με διάφορα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι ο προβληματισμός αυτός ε, απεικονίζεται και στο σχέδιο που παρουσίασα στο Συμβούλιο. Ε, θέλω έναν ειδικό εκπρόσωπο ο οποίος θα υλοποιήσει τις βασικές μας προτεραιότητες, θα προωθήσει τα θέματα τα οποία πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Σαλαφράγκα, η κατάργηση της αρνητικής ποινής, ε, καταπολέμηση της χρήσης των βασανιστήριων, προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, των παιδιών, να και για να τα εξασφαλίσουμε όλα αυτά, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνεργαστούμε μεταξύ μας και βεβαίως με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η θητεία αντί για ένα χρόνο θα είναι διετής, μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διορίσει έναν ειδικό αντιταλμένο για ειδικά θέματα, με θεματική εντολή δηλαδή. Θα πρέπει λοιπόν ε, να του δώσουμε μια εντολή αρκετά μεγάλη ε, χρονικά, ούτω ώστε να εξασφαλίσει αυτά, να προωθήσει αυτά τα θέματα. Ο δικό ε, εκπρόσωπο πρέπει να έχει εμπειρία και πραγματογνωμοσύνη για να και θα πρέπει να έχει πραγματική εμπειρία και κατανόηση από ανθρώπινα δικαιώματα και από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τα κράτη-μέλη έχουν ε, προτείνει κάποιους θαυμάσους υποψηφίους και θέλουμε να προωθήσουμε γρήγορα αυτόν τον διορισμό. Θέλω να ξεκαθαρίσω όμως ότι ο ειδικό εκπρόσωπο θα είναι σημαντικό συνομιλητή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε την ε, δέσμευσή μου ότι όποιο και αν είναι αυτό ή αυτή θα ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τακτικά ε, με βάση τις ε, που θα έχουμε κανονίσει. Επίσης θα, θα προσθέσει ε, προσθέμενη αξία στη δουλειά μας και θα είναι ηγηθή των, του διαλόγου και των διαβουλεύσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. θα είναι ο φυσικός συνομιλητής και εταίρος. Η... Επίσης η διπλωματία και τα επικοινωνιακά θέματα θα είναι πολύ βασικά. Θα πρέπει να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά για να το ξεκαθαρίσω, ε, και εγώ προσωπικά θα παραμείνω, θα εγγύψω επί, του θέματος και θα με βοηθήσει και η ομάδα μου στις Βρυξέλλες αλλά και στο εξωτερικό τους. Ε, ευχαριστώ σήμερα ε, για τη δουλειά που κάνουν τα τελευταία χρόνια. Και Φυσικά, αυτό είναι τμήμα ενό μεγάλου πακέτου. Ε, θα υιοθετηθεί τώρα το στρατηγικό πλαίσιο για την εξωτερική δράση ε, και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι τμήμα αυτή. Με βάση τις δεσμεύσεις που έχω λάβει θα σας ε, εμπλέξω και εσά σε αυτή τη διαδικασία. Είναι τελευταία συζήτηση από μια σειρά συζητήσεων που έχουν γίνει για αυτό το θέμα κυρία Λοχμπίερ ήταν πρόεδρος αυτών των επαφών ε, με τις οποίες ε, η υπηρεσία μου ήρθε σε, επαφή και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια πιο πλήρη και ευρεία προσέγγιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Θέλω να έχουμε μια ευρεία προσέγγιση και να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ε, ενδιαφερόμενους, όλους τους stakeholders να συνεισφέρουν για να διαμορφώσουμε την πολιτική μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Σαλαφράγκα ακόμα μια φορά για την εκθεσή του. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος ε, Πρέντα για 1,5 λεπτό από τις πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ η συνθήκη είναι σαφής. Η Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αξίες ε, βάσει των οποίων εδραιώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Η κυρία Άστον ξεκίνησε διακηρύσσοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αποτελέσουν το πυρήνα της εξωτερικής της πολιτικής και η δράση μέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν εναρμονιστεί. Και αυτό στο παρελθόν έχει ε, κατακριθεί ε, αν ε, καθορίσουμε έναν εντεταλμένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα να γνωρίσουμε την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στον τομέα αυτό και από την άλλη πλευρά εάν θεωρήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σαν έναν ειδικό τομέα εάν τα λαμβάνουμε υπόψη μας μόνο στις συγκεκριμένες συζητήσεις και όχι στις γενικές συζητήσεις με τους αρχηγούς κρατών δεν νομίζω ότι θα επιτύχουμε το στόχο μας διότι η Αραβική Άνοιξη μας υπενθύμησε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια και ο ένας πρέπει να μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινά του δικαιώματα και να μπορεί να λειτουργεί ε, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα κράτη να βασίσουν τη δραστηριότητά τους εις, ε, του, εις, ε, εις, τις αρχές. Δεν βλέπω τον κύριο Χάουιτ και δίνω το το λόγο τώρα στον κύριο Ντόνσκης για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ο καθορισμός ενός επιτετραμένου για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι στρατηγική απόφαση και ελπίζουμε ότι μια τέτοια θέση θα μπορέσει να εξασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα έχουν ακόμη πιο εξέχουσα θέση στη δράση μας και θα προωθηθούν. Θα ελπίζουμε ότι το άτομο αυτό θα βρει την σωστή του θέση στο περιβάλλον περιβάλλον στο οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει και θα πρέπει να επέμβει αμέσως. Ελπίζω δε ότι θα καθορίσει προτεραιότητες που πρέπει να επιληθούν και θέλω να τονίσω εδώ ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει την πολιτική μου ομάδα και πρέπει να αποφευθούν οι αυτοπυρπολισμοί των μοναχών και ε, να μπορέσουμε να εξετάσουμε αν χρειάζεται ένας ειδικό εντεταλμένος για το Θιβέτ και μόνο. Ε, όσον αφορά τα εντεταλμένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί μόνο μία πτυχή της στρατηγικής μας για να επιδείξουμε την πολιτική μας βούληση να ενισχύσουμε την συνεργασία μας στον τομέα αυτό επί του διεθνούς επίπεδου και επιπλέον να υπάρχει ένα διαθεσμικό έγγραφο, μία φιλόδοξη διακήρυξη όπως η Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη όπου τα κράτη-μέλη αναπτύσσουν την πολιτική τους. Να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μία συνένεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο με συγκεκριμένες ενέργειες για να επιτύχουμε τους στόχους μας γιατί μόνο έτσι θα επιτύχουμε και προσβλέπω στην συνεργασία επί του θέματος στην Ευρώπη. Τον λόγο έχει τώρα ο κύριος Σταβάρες για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία είπατε εκπρόσωπε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολλά χρόνια τάχθηκε υπέρ ε, της, του διορισμού ενός ειδικού εντεταλμένου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ και χρόνια ε, απευθύναμε έκκληση για το διορισμό αυτό. Βρισκόμαστε στα τελευταία μέτρα αυτού του μαραθώνιου. Δύο στοιχεία μας λείπουν για να είμαστε βέβαιοι ότι όλα θα πάνε καλά με το διορισμό του νέου ειδικού εντεταλμένου. Θέλουμε έναν άνθρωπο που θα είναι κατάλληλος ε, για τον πρώτο καιρό, για να γίνει αυτό το πρόσωπο του ειδικού εντεταλμένου κατά την πρώτη αυτή φάση της ανάλυσης των καθηκόντων και όπως είπε και ο συγητής ε, Σαλαφράγκα θα πρέπει να έχει στενή συνεργασία με, την, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να προσδιορίσουμε με σαφήνεια την εντολή του. Θα πρέπει φυσικά αυτός ο, ο άνθρωπος να μην δημιούργησε ένα γκέτο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αντίθετα να αποτελεί έκφραση όλων των πολιτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω όλων των πολιτικών της Ένωσης, των εμπορικών συμφωνιών, των διμερών συμφωνιών με χώρες, με πολυμερών συμφωνιών με ομάδες χωρών και επίση να επικεντρωθεί σε κάτι πολύ σημαντικό για το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουμε, σε αυτά τα τελευταία μέτρα στην τελική ευθεία αυτού του μαραθωνίου. Δεν καταλαβαίνω γιατί είπα ότι εκπρόσωπος που είναι είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτός ο ειδικό εντεταλμένο δεν περιλαμβάνει ακόμη στην εντολή του και θα ήθελα μία απάντηση οριστική για αυτή την εντολή. Δεν έχει την ε, ε, αυστηρή ευθύνη λογοδοσία απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να είναι ειδικό εντεταλμένο τη Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί ρητή και κατηγορηματική ευθύνη λογοδοσία απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε ε, τον ειδικό εντεταλμένο εδώ, στη συζήτηση των κατεπηγόντων στο Στρασβούργο και θέλουμε επαφή με την ομάδα επαφή και στενή συνεργασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, αυτή η ομάδα θα θεσμοθετηθεί, θα επισημοποιηθεί και θα έχει συγκεκριμένο ρόλο. Ευχαριστώ που είπατε ότι είστε υπέρ των επαφών με την ομάδα εργασίας, αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο και για αυτό το σημείο. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στον κύριο Χόουιτ που έχει καταφτάσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, με συγχωρείτε που καθυστέρησα, αλλά θέλω να χαιρετήσω την διαβεβαίωση ε, ε, ε, της είπα της εκπροσώπου ότι θα καθοριστεί ένας ειδικό εκπρόσωπος, διότι θα είναι ένας επιτετραμένος στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφαλείας που θα αποδειξεί ότι δίνουμε το σωστό, τη σωστή σημασία στο βασικό αυτό θέμα και θα ενισχύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με ε, τον προηγούμενο προσωπικό εκπρόσωπο ενώ τώρα θα είναι ένας εκπρόσωπος εν ονόματι ε, της ΥΠΑ του εκπροσώπου αλλά σε συνεργασία με το Συμβούλιο και ελπίζω και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι αυτά τα οποία έχουν λεχθεί στο ψήφισμα και στις συζητήσεις που έχουν ήδη ήδη γίνει ε, σας πείθουν ότι χρειάζεται ένας ε, υψηλού επίπεδου εκπρόσωπος της υπάτου εκπροσώπου κατά τρόπον ώστε να μπορεί να συμμετέχει και στις συζητήσεις στο ε, ε, Διεθνές ε, Ποινικό Δικαστήριο και θα μας ενισχύσει τη θέση μας σε σχέση με το παρελθόν. Κάτι το οποίο για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάρα πολύ βασικό στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία να πετύχουμε το στόχο μας και γι' αυτό επαναλαμβάνω στην ύπατη εκπρόσωπο ότι δεν θέλω αυτό να είναι μία απλώς πολιτική, ένας πολιτικός καθορισμός αλλά ένα άτομο το οποίο θα εφαρμόζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, παρόλο που είναι κάποιος που θα επιλεγεί αποκλειστικά και μόνο από την ύπατη εκπρόσωπο ε, θα πρέπει να είναι ένα άτομο το οποίο θα έχει ήδη ένα παρελθόν ε, και δείγματα γραφής στον τομέα αυτό κατά τρόπον ώστε να αποδειχθεί ότι είναι μια μεγάλη προτεραιότητα. Υπάρχει μια μπλε κάρτα την οποία σας ε, δίνει ο κύριος Ντάρτμουθ. Ε, την δέχεστε κύριε Χάουιτ. Κύριε Χάουιτ. Είσαστε υπέρ του διορισμού από ό,τι φαίνεται ή μάλλον υπέρ των πολιτικών διορισμών. Μήπως ε, και ο ίδιος ο διορισμός της ίδιας της ΥΠΑ του εκπροσώπου ήταν πολιτικός. Τι λέτε, δεν ήταν ή ήταν. Δεν ξέρω αν ακούσατε το λόγο μου. Εγώ ήμουν κατά των πολιτικών διορισμών. Μάλλον δεν ακούσατε καθόλου την ομιλία μου. Το λόγο έχει ο κύριος Μπιέλλαν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν μία από τι υποχρεώσει που αναλάβαμε ω Ευρωβουλευτέ. Πραγματοποιώντα την πολιτική συνεργασία με πολλέ χώρε, πολύ συχνά συναντάμε διάφορε εκφάσει αυτού του προβλήματο τη ε, διάκριση ε, ει βάρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδιαίτερη σημασία έχει αυτό το θέμα σε σχέσεις με, στεν... με σημαντικούς γειτονές μας ή χώρες με ενταξιακές βλέψεις. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως στις χώρες που έχουν άμεση σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Λευκορωσία, εδώ και πολλά χρόνια από αυταρχικό καθεστώς που με βίο τρόπο καταστρατηγεί τα δικαιώματα και εξολοθρεύει πολιτικού αντιπάλου. Σε πολλέ ε, χώρε τη πρώην Σοβιετική Ένωση έχουμε τέτοιε συμπεριφορέ ε, που καταστρατηγούν τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα στη, πιο συχνά πρόκειται για απομεινάρια της προηγούμενης εποχής και έχουμε πολλές φορές ε, και, κακή, και κατάχρηση της εξουσίας από δημοκρατικά εκλεγμένες εξουσίες. Λοιπόν, θα πρέπει με τις δράσεις μας να αναβαθμίσουμε τις πολιτικές προδιαγραφές στις χώρες αυτές και αυτό είναι μια σημαντική υποχρέωση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Θα πρέπει λοιπόν με τον διορισμό του ειδικού εντετελμένου διευκολύνουμε την κατάσταση αυτή, αλλά θα πρέπει να έχει στενή συνεργασία με την έπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική και να βρίσκεται φυσικά υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Αυτό είναι απαραίτητη προπόθεση για να εξασφαλίσουμε τη συνοχή τη εξωτερική μα πολιτική. Θα ήθελα εν κατακλείδη να τονίσω ότι η πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο θα πρέπει να συνδυαστεί με το σεβασμό των παραδοσιακών δικαιωμάτων τη οικογένεια και παρόμοιων αξιών. Για παράδειγμα, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών, ακόμη και αυτών που, δια, που διαπράττονται στο όνομα εσφαλμένη αντίληψη θρησκευτική ουσία ορισμένων λατριών. Ευχαριστώ. Το λόγο κύριο Ντάρτμουθ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ανθρώπινα δικαιώματα ή όχι ανθρώπινα δικαιώματα. Θα παίρνετε, θα έχετε, θα πληρώνετε 12 εβδομάδε για διακοπές, πληρωμένες διακοπές, δηλαδή κάτι που συμβαίνει γενικά στην εξωτερική υπηρεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, εμείς ε, έχουμε υποτίθεται ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ιερά και απαραβίαστα. Α, όμως τι λέμε για τα θύματα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Ε, υπάρχουν Βρετανοί υπήκοοι ε, που χάρη σε αυτό το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη ε, κρατήθηκαν στην Ελλάδα και μάλιστα κρατήθηκαν στη φυλακή του Κορυδαλού. Απλώς πιάσαν, είχαν πιάσει οι Έλληνες λάθος άνθρωπο και το βάλαν στη φυλακή αυτή για μήνες. Διάφοροι Βρετανοί υπήκοοι έχουν κλειστεί σε φυλακές της Ευρώπης και εμείς λοιπόν είμαστε θύματα και έχουμε προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, θα πρέπει πρώτα εμείς να τακτοποιήσουμε τα του οίκο μας πριν να αρχίσουμε να χώνουμε τη μύτη μας και αλλού. Ε, σε τι κατάσταση δηλαδή ε, είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εξωτερικό. Ε, το Μάρτιο του 2010 η ύπατη εκπρόσωπος ε, γίνει πολλά μάλλον το 2010 και μετά, αλλά η ύπατη εκπρόσωπος δεν έχει μάθει τίποτα. Δεν έχει διδαχθεί από το παρελθόν. Η κυρία Σανκλέρ. Ευχαριστώ. Ε, κύριε, ο συνάδελφος θα ήθελα να μας πει πώς, ε, τι άποψη έχει για αυτά που είπε ο προλαλής σας. Γιατί δεν απαντήσατε τις ερωτήσεις του. Αν έχουμε αξιοπιστία, θα πρέπει να σεβόμαστε την ε, μπλε κάρτα. Γιατί σας ρώτησα και κάτι άλλο. Σας είπε, δεν σας είπε μόνο τι πιστεύετε για τους πολιτικούς διορισμού, αλλά τι πιστεύετε και για τον πολιτικό διορισμό της κυρίας Άστον. Παρακαλώ απαντήστε λοιπόν σε αυτή την ερώτηση που σα έκανε ο προηγούμενος Ευρωβουλευτής, κύριε Χάουιτ. Θα διαπιστώνω ότι α, ανησυχείτε πολύ για τις εργασιακές συνθήκες του ειδικού εντεταλμένου, ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σας αφήνω λίγο χρόνο να βάλετε τα ακουστικά σας. Λοιπόν, βλέπω ότι ασχολείστε ιδιαίτερα με τις εργασιακές συνθήκες του ειδικού εντεταλμένου. Θα ήθελα να πω, α, αντί να ασχολείστε με το θέμα αυτό, δεν θα πρέπει να μας πείτε αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι στην εντολή του δεν περιλαμβάνεται υποχρεωτική λογοδοσία απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι ε, είναι πολύ πιο σημαντικό να έχει λογοδοσία απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρά να δικαιολογεί τι συνθήκε εργασία και άδειά του. Η ερώτηση τη κυρία Σενκλέρ δεν ήταν ερώτηση προς τον κύριο Χόιτ, ήταν μάλλον διαπίστωση. Κύριε Ντάρτιν, θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Ταβάρε. Για αυτό που κυρία, ε, η κυρία Σίνκλερ. Μάλλον κύριε Χάουιτ, ε, θεωρείτε ότι εσάς δεν σας καλύπτουν οι κανόνες περί ευγένειας. Για αυτά που είπε ο κύριος Ταβάρες. Μάλλον εγώ με τον κύριο Ταβάρες ε, δεν συμφωνούμε για τα περισσότερα πολιτικά θέματα. Αλλά κύριε Ταβάρε, ίσως σας εκπλήξει το γεγονός ότι εγώ συμφωνώ, αν αυτό είπατε, εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία, ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Το πρόβλημα είναι ότι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε άλλο. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Με αυτό λοιπόν έχουμε αντίρρηση. Όχι με τίποτα άλλο. Κύριε Χάουιτ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ε, θα ήθελα να είμαι καταρχήν ευγενής προς όλους οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες και όχι από το Ενωμένο Βασίλειο και οι οποίοι θα βαριούνται μέχρι δακρύων για αυτή την εσωτερική διαφωνία. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Χατζηγεωργίου για ένα λεπτό. Κύριε Χατζηγεωργίου, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ο διορισμό ειδικού εντεταλμένου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί και πρέπει να αποβεί μια ωφέλιμη εξέλιξη, εφόσον βέβαια τηρηθούν κάποιε κατευθύνσει. Το κυριότερο απ' όλα είναι η λογοδοσία στην οποία θα υπόκειται απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά δεύτερον, εναπόκειται στην ελευθερία δράση που θα έχει ο συγκεκριμένο άνθρωπο ή πολύ περισσότερο η ελευθερία που θα κατακτήσει κατά την υλοποίηση των καθηκόντων του η ευρωπαϊκή ένωση μπορεί και πρέπει να αναδείξει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ζήτημα κρίσιμης σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας. για να επιτευχθεί όμως αυτό χρειάζεται βαθιά πίστη ότι οι πολιτικέ σκοπιμότητες, και το υπογραμμίζω αυτό δεν θα έχουν λόγο και ρόλο στην δραστηριότητα του συγκεκριμένου εντεταλμένου γύρω από το ζωτικό ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. έχει επίση τεράστια σημασία ποιο θα αναλάβει αυτό το πόστο πόσο υπόλογο θα είναι σε αυτού που θα τον διορίσουν πόσο υπόλογο θα είναι όπω είπα πριν και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και σε ποιο βαθμό θα αντιλαμβάνεται ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να τύχουν σεβασμό σε κάθε σημείο του κόσμου αλλά και στην ίδια την ευρωπαϊκή ένωση. κλείνω λέγοντα ότι διαρωτούμε αν ο συγκεκριμένο αντιπρόσωπο θα έχει δικαίωμα ή υποχρέωση να δει την βάναυση παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κράτη μέλη τη ευρωπαϊκή ένωση από χώρε που έχουν αιτηθεί την ένταξή του στην ένωση. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Σανκλέρ για 1,5 λεπτό. Καταρχήν κυρία Πρόεδρο, ο έκανα μία ερώτηση. Αν κάποιος συνάδελφο συμφωνεί μαζί μου είναι ερώτηση και θα έπρεπε να λάβω απάντηση. Αλλά ε, το 1976 ε, είχαμε θεσμοποιήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και στη χώρα μου, στη Μεγάλη Βρετανία, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι της αρμοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά αυτό δεν αρκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητήθηκε ένας ειδικό εκπρόσωπο ε, με προσωπικό και γραμμή του προπολογισμού για το συγκεκριμένο θέμα. Κυρία Σενκλέρ, μπορείτε να μιλήσετε λίγο πιο αργά, διότι οι διερμηνείς δεν προλαβαίνουν. Με, ε, με διακόψατε, μπορώ να ξεκινήσω από την αρχή μπορείτε να συνεχίσετε. Έχουν μεταφράσει, αλλά για τη συνέχεια μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά. Με συγχωρείτε, αλλά δεν ξέρω που βρίσκομαι τώρα. Μπορώ να ξεκινήσω από την αρχή και να μιλήσω πιο αργά, γιατί δεν ξέρω που βρισκόμουν. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά ξεκινήστε. Το 1776 ε, ο Τόμας Τζέφερζον περιείχε τα ανθρώπινα δικαιώματα στη διακήρυξή του και τώρα πρέπει να τα προστατεύουμε όπου και να βρισκόμαστε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι της αρμοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά αυτό δεν αρκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο εισηγητής ζητά να υπάρχει ένας ειδικό εκπρόσωπος με προπολογισμό και προσωπικό και ε, αυτή η αντιπροσωπεία θα έπρεπε να είναι πιο υπεύθυνη ε, διότι ε, πέραν, των δικαιωμάτων για αργίες και διακοπές έχουμε 119 τέτοιες αντιπροσωπείες και αυτό το οποίο συμφωνώ στην έκθεση είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε έναν εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που να γνωρίζει το θέμα και να μπορέσει να τα προασπίσει και να έχει και διεθνές κύρος. Αυτά τα κριτήρια βέβαια δεν είχαν ληφθεί υπόψη όταν καθορίστηκε η ύπατη εκπρόσωπος. Ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Κούκαν για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ θερμότατα τον εισηγητή μας για το πολύ αξιόλογο έργο του στην έκθεση αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τώρα μία ευκαιρία με την έκθεση αυτή και τη σύστασή του να συμβάλλει στη συζήτηση προκειμένου να διαμορφωθεί ο ρόλος και η θέση του ειδικού εντεταλμένου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Κοινοβούλιο για πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό στη σύστασή μας κάνουμε πολλές εκκλήσει και συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγγνώμη, και ελπίζω να γίνουν δεκτές. Πρώτα απ' όλα, ο ειδικό εντεταλμένο θα πρέπει να έχει μια ανεξάρτητη και ελαστική εντολή, ώστε να μπορεί να ενεργεί άμεσα και αποτελεσματικά. Θα πρέπει ο ειδικό αυτό εντεταλμένο να ε, βελτιώσει και να ε, ενισχύσει την προβολή και την ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τα θέματα ε, πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει συνοχή και mainstreaming το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την οριζόντια λήψη υπόψη σε όλες τις πολιτικές υπόψεις, ε, σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Θα πρέπει να γίνει υψηλός, υψηλό επίπεδο διαμεσολαβητής με τους εταίρους μας, στις τρίτες χώρες και με τις διεθνείς οργανώσεις. Θα πρέπει να μας εκπροσωπεί σε διεθνή φόρα και να έχει σχέσεις και με τον ΟΗΕ και με διάφορες περιφερειακές ε, οργανώσεις. Θα ήθελα τέλος να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πολύ ευχαρίστω θα συμμετέχει στη διαδικασία διορισμού και ιδιαίτερα στην ακρόαση που θα έχουμε με τον υποψήφιο ή την υποψήφιο και επίσης θα θέλαμε να επιβλέπουμε και την εντολή καθ' όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σενίσιν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ παρά τις μέχρι τώρα προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της είπε της εκπροσώπου της κυρίας Άστον, την οποία ευχαριστούμε θερμά, ε, δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της τυπικής κατοχήρωσης και της ουσιαστικής εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήδη στην έκθεση του κυρίου Χόουιτ λέμε ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι όχι μόνο συνεπής, αλλά θα πρέπει να είναι και υποδειγματική. Ο διορισμός του ειδικού εντεταλμένου της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενισχύει τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την ελευθερία, και τη θέση των ακτιβιστών υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εντολή και τι αρμοδιότητέ του θα πρέπει να αντανακλά την πολιτική τη Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα η, κατά, η κατάργηση τη θανατική ποινή, ο περιορισμό των καταπολέμηση των βασανιστήριων, η, η πάταξη των διακριτικών μεταχειρήσεων κατά των γυναικών, των LGBT, η ελευθερία έκφρασης και στο διαδίκτυο, η ανεξιθρησκεία, ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες και ούτω καθεξής. Ε, έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον κόσμο των επιχειρήσεων. Γι' αυτό συμφωνώ με τη διεύρυνση της εντολής ε, ως προς αυτή την κατεύθυνση του ειδικού εντεταλμένου και την επέκταση των συστάσεων και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΗΕ ό,τι αφορά την επέκταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στι επιχειρήσει. Θα πρέπει να συνεργάζεται ο ειδικό εντετελμένο με τον ΟΗΕ και με την ομάδα εργασία του ε, Συμβουλίου, καθώ και με περιφερειακέ οργανώσει ή με εμπειρογνώμονε και άλλε οργανώσει που προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μεταξύ των υποχρεώσεών του θα πρέπει να είναι μια ανεξάρτητη και ελαστική εντολή και φυσικά θα πρέπει να εφοδιαστεί με τα απαραίτητα μέσα για να διεξαγάγει το έργο του. Θα πρέπει φυσικά το πρόσωπο αυτό να έχει ιδιαίτερα προσόντα, δεξιότητες, κύρος στο παγκόσμιο προσκήνιο, πλούσια πείρα, να έχει εμπειρογνωμοσύνη ε, σε θέματα ανθρωπιστικού δικαιωμάτου, αλλά και σε θέματα απονομής ε, διεθνούς δικαιοσύνης. Ευχαριστώ κυρία Σενίση, η κυρία Λόχ Μπίλερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και κυρία Ήπατη εκπρόσωπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περιοχή η οποία θέλει να προωθήσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενεργά και γι' αυτό πρέπει να έχουμε έναν ειδικό απεσταλμένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θα είναι εύκολη δουλειά για να υπάρξει μία θέση είτε διμερής είτε πολυμερής και η οποία θα υιοθετηθεί και δεν θα πρέπει κανείς να υποθάλπει την πολιτική αυτή αλλά να τη στηρίζει επικοδομιακά ε, ε, επικοδομητικά. Προηγουμένως ε, είχαμε αναφέρει ότι χρειάζεται μία καλύτερη πολιτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρακολουθούμε και στηρίζουμε και θα στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Ο ειδικό εντεταλμένος θα πρέπει να μπορεί να ενημερώνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ θα ήθελα αυτό να διατυπώνεται πρόσαφώς κατά τρόπον ώστε η εισηγητής ή η εισηγήτρια να είναι ενημερωμένος ε, συχνά κατά τρόπον ώστε να μπορέσει να ικανοποιηθεί αυτή η προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τέλος σας εύχομαι ε, καλή επιτυχία στην επιλογή ε, του ειδικού εντεταλμένου. Χρειαζόμαστε ε, ένα άτομο κύρους με γνώσεις και επιμονή που θα μπορέσει να επιβληθεί επί σειρά ετών στο έργο αυτό. Ο κύριος Βαντάλεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. ο διορισμό ενό ειδικού εντεταλμένου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μα δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε περισσότερη προσοχή στο θέμα αυτό, στα ανθρώπινα δικαιώματα δηλαδή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά που συχνά αγνοείται και παραβλέπεται. Η θρησκευτική ελευθερία είναι μια από τι πιο σημαντικέ ελευθερίε. Έχουμε εξτρεμιστέ μουσουλμάνου, οι οποίοι επιτίθενται σε χριστιανού ορισμένε χώρε. Φερρυπίν. Κάθε εβδομάδα σε ορισμένε χώρε σκάνε βόμβες σε εκκλησίες. Πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να δώσουμε μεγάλη σημασία και στην θρησκευτική ελευθερία. Ο ειδικό αυτός εκπρόσωπος είναι και μια νέα ευκαιρία για μας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πώς εφαρμόζονται και στην Ευρώπη και αλλού. Στην Ινδία υπάρχουν χιλιάδες άτομα τα οποία ε, σκλαβώνονται. Δεν μπορούμε να έχουμε εμπορικέ συμφωνίε ε, με κάποιε χώρε χωρί να έχουμε και μία ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επόμενο ομιλητή για 1,5 λεπτό. Ο κύριο Γκζιμπ. Ευχαριστώ. Η σημερινή συζήτηση δεν είναι μία σκέψη που ξεκίνησε παρασκηνιακά, ιδιωτικά ε, αλλά είναι πολύ σημαντική συζήτηση επευκαιρία ευκαιρία της σύστασης προς το Συμβούλιο και απορρέει από το άρθρο 28 τη ε, Συνθήκη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλάει για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και των θεμελιωδών δικαιολευθεριών, καθώ και από το άρθρο 33 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλάει για το διορισμό ειδικού εντεταλμένου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίση αυτή η συζήτηση είναι απόρρια και διάφορων διεθνών συζητήσεων όπως το Δεκεμβρίου του 2011 για την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Το αποτέλεσμα λοιπόν επίσης το σκέψεων και το συζητήσω μετά από τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης. Ο διορισμό του ειδικού εντεταλμένου θα πρέπει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την προβολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μα λείπει πολλέ φορέ η συνοχή τη κοινοτική πολιτική στα θέματα αυτά. Και επίση θα πρέπει να έχει ιδιαίτερο ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο διορισμό και στην επίβλεψη των εργασιών και των δραστηριοτήτων του ειδικού εντεταλμένου θα πρέπει επίσης να γίνει σημαντικός διαμεσολαβητής υψηλού επίπεδου με τρίτες χώρες, με διεθνείς οργανώσεις, με περιφερειακές οργανώσεις και ούτω καθεξής. Ο μελλοντικό αυτός ειδικό συντεταλμένο, θα πρέπει να είναι άνθρωπος με ιδιαίτερο κύρο στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ των οργανώσεων και των θεσμικών οργάνων και να είναι γνωστός γιατί θα εγγυηθεί μια πραγματική και κατάλληλη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους εταίρους στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το λόγο κύριο Λάιχτφριντ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Ήπατη εκπρόσωπο. Πιστεύω ότι μπορούμε να συζητάμε για την ευρωπαϊκή πολιτική και να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά πρέπει να πούμε ότι πάντοτε η ευρωπαϊκή πολιτική έχει επιδείξει ε, ένα σταθερό σημείο που είναι η θέλησή της για επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι καλό αν αυτή τη στιγμή στιγμή καθορίζεται ένας ειδικό εντεταλμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό και μόνο το θέμα. Δεν πρόκειται ε, παρά για ένα καλό θέμα και καλό δείγμα. Πρέπει βέβαια να τον ρωτήσουμε τι είναι σε θέση να κάνει και από εκεί και πέρα θα δούμε. Αυτό που είναι βασικό είναι να έχει μία ευρεία εντολή, να μην είναι περιορισμένη η εντολή του να μην πρόκειται ε, για τα τετριμένα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά να μπορεί αυτός να αποφασίσει σε ποια θέματα θα αφιερωθεί να έχει μία εντολή αρκετά μακρά και πιστεύω ότι ε, θα πρέπει ε, να είναι τουλάχιστον δυόμιση χρόνια δηλαδή το ίμιση της θητείας του Ευρωκοινοβουλίου και επιπλέον χρειάζεται να είναι μία να υπάρχει σωστή επάνδρωση και το αναγκαίο προσωπικό. Αυτό που εμένα θα με ενδιαφέρε είναι να, μπορεί να αποδίδει λογαριασμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να είναι υποχρέωσή του αυτό ε, γιατί πρέπει να ελέγχουμε τι κάνει και τι γίνεται. Ένα άλλο που με ενδιαφέρει και τελειώνω είναι ότι δεν πρόκειται για πολύ ευραία θέματα αλλά παραδείγματος να μπορεί ε, να παρακολουθήσει παραδείγματο χάρη τι κάνουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεω στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, εγώ ήθελα να σχολιάσω και κάτι στον Earl of Dartmouth αλλά έφυγε και έτσι τελειώνω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιγκάλσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η πρόσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, θα πρέπει να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να εξασφαλίσουμε την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εντό Ευρωπαϊκή Επικράτεια, αλλά και σε όλε τι χώρε με τι οποίε συνεργαζόμαστε και, στις οποίες, ε, και για την εσωτερική κατάσταση των οποίων έχουμε κάποια επιρροή. Είναι σημαντική αυτή η έκθεση και αυτή η σύσταση. Βέβαια υπάρχουν κάποια σημεία που είναι λίγο ανησυχητικά σε ό,τι αφορά ε, την ε, ε, σύγχυση που γίνεται μεταξύ της σεξουαλικής ελευθερίας και της πάταξης των βασανιστήριων. Πέραν αυτών των αμφιβολιών και τη δική μου αντίληψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η λειτουργία και πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη σύσταση και την έκθεση για το διορισμό του ειδικού εντεταλμένου, γιατί η δημιουργία αυτής της θέσης είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι ο διορισμός αυτός θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλους. Ευχαριστώ κυρία Γέγκλε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Άστον, καταρχήν σας ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική έκθεσή του, διότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει ε, να αντικατοπτρίζεται σε όλους τους τομείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ιδίως στο αυτόν τον ευαίσθητο τομέα είναι απαραίτητο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη να μιλούν με μία φωνή και να έχουν μία συνεκτική και υπεύθυνη δράση. Γι' αυτό και εδώ και πολύ καιρό έχουμε ζητήσει να υπάρξει ένας ειδικό επιτετραμένος Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτή η επιτετραμένη δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ένα συγκεκριμένο θεματικό τομέα, αλλά θα πρέπει να δρούν υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να παρακολουθούν ότι υπάρχει εφαρμογή του κράτους δικαίου. Αυτό πρέπει να συμβαίνει και στη συνεργασία του ειδικού επιδετραμένου με άλλους υψηλά ισταμένους και θα χρειάζεται να μπορεί να συνεργαστεί με πολιτικά υπεύθυνα άτομα αλλά και με την κοινωνία των πολιτών σε όλα τα επίπεδα όπως άλλωστε και στη, με εθνικές και διεθνείς οργανώσεις. Μόνο αν υπάρχει στενή εμπλοκή της τοπικής της κοινωνίας και της ε, εθνικής θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση κατά τρόπον ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει και αυτό να καλύψει τον ρόλο του και να παρακολουθεί τη δράση του εντεταλμένου αυτού γι' αυτό και ελπίζω ότι ο κύριος αυτός θα έρχεται τακτικά να μας ενημερώνει για τις δραστηριότητες του. Ευχαριστώ στην κυρία Γκέγκλη, κυρία Γκόμης για δύο λεπτά. Ο διορισμό ενό εντεταλμένου μια εντεταλμένη για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αποτελεί πρόοδο τη ευρωπαϊκή πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι θεμελιώδει ε, ελευθερίε. Και όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά οικουμενικό και καθολικό όλοι οι εντεταλμένοι θα πρέπει να έχουν πολιτική πείρα, σημαντικά διαπιστευτήρια στα θέματα ανθρωπιστικού δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώματα, σε θέματα διεθνού δικαιοσύνη και επίση ε, να μπορεί ο άνθρωπο αυτό ε, να είναι στρατηγικό και ευφύ συνήγορο υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Θα πρέπει να μιλά εκ μέρου Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, να έρχεται και να λογοδοτεί όποτε είναι απαραίτητο και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει ο ειδικό αυτό εντεταλμένο να εξασφαλίσει την εφαρμογή κατευθυντηρίων γραμμών και ε, διαφόρων σχεδίων δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει θαραλέα και τολμηρά να ε, στιγματίζει καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε χώρα με την οποία έχουμε έστω και προνομιακές σχέσεις. Θα πρέπει να είναι θαραλέος και να στυλιτεύει τέτοιου είδους παραβιάσεις. Επίσης θα πρέπει ε, να να αποφύγουμε εμπορικές συμφωνίε ή οικονομική στήριξη σε αυταρχικά καθεστώτα που καταστρατηγούν τα δικαιώματα των λαών τους. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στις χώρες εταίρους μας και να προαγάγουμε τα δικαιώματα τη κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι προτεραιότητα τη εξωτερική μα δράση. και η στρατηγική ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι σε κάθε χώρα θα πρέπει να διαμορφώνεται από κοινού με την κοινωνία των πολιτών και οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να δημοσιεύονται. Ελπίζω το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν και να εξασφαλίσουν μια απόλυτη συνεργασία με το αντίνατεταλμένο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διευκολύνουν το έργο συντονισμού ε, και ε, για τις ε, λειτουργίες που θα κληθεί να αναλάβει. Ελπίζω ότι θα κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή, κυρία ήπατε εκπρόσωπε. Κυρία Γκάλ, για ένα μισή λεπτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Επιτέλους η θέση του ειδικού εντεταλμένου θα δημιουργηθεί και ελπίζουμε γρήγορα να πληρωθεί. Ελπίζω να μην ε, γίνει απλώς, δημιουργηθεί απλώς μία θέση, αλλά ένας ολόκληρος φορέας, ένας ε, θεσμός. Εμείς ε, προωθούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το σεβασμό των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα σχέδια συμπερασμάτων των Συμβουλίων μιλούν για τη διετία αυτή που γιατί η αρχική πρόταση του Κοινοβουλίου ε, είχε ζητήσει να επεκτείνουμε την ε, εντολή του ειδικού εντεταλμένου. Θα χρειαστεί εξάλλου και χρόνος για να δημιουργηθεί ας πούμε, μια υπηρεσία. Πρέπει το, η εντολή αυτή να είναι κατάλληλη, να είναι ευέλικτη και να δοθούν επαρκείς πόροι, ούτω ώστε να προσδιορίσουμε το σωστό τρόπο την ε, εντολή αυτή. Επίσης, ο ειδικό αντεταλμένο εκπρόσωπο θα πρέπει να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να δούμε κατά πόσον ε, υλοποιεί σωστά την εντολή του. Με αυτή τη θέση κάνουμε ακόμα ένα βήμα, ούτω ώστε να έχουμε μια πιο αποτελεσματική στρατηγική ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Κύριε Κοπά. Ο βασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί τον πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά με τη δημιουργία της θέσης του ειδικού εντεταλμένου της ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. ζούμε σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών σε πολλές χώρες με τις οποίες η ένωση θέλει να διατηρεί καλές σχέσεις. άρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να προστατεύονται και να προβάλλονται οι αξίες μας που είναι ο σεβασμός του ανθρώπου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας η ελευθερία η ισότητα και η αλληλεγγύη ο διορισμός του ειδικού εντεταλμένου θα βοηθήσει έτσι ώστε η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να γίνει πιο αποτελεσματική στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επειδή ο ειδικός εντεταλμένος θα μπορεί να δρά γρήγορα και άμεσα. είναι επομένως απαραίτητο να του δοθεί ξεκάθαρη εντολή για το πεδίο δράσης για να μην δημιουργείται σύγχυση ανάμεσα στις σχετικές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων για το ποιος είναι αρμόδιος επίση η χρονική διάρκεια του διορισμού είναι απαραίτητο να μπορεί να επιμεκυνθεί εφόσον ο ειδικό εντεταλμένο αποδείξει την επάρκειά του. το πρόσωπο που θα επιλεγεί πρέπει να έχει αποδείξει έμπρακτα με τη δράση του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι έχει τι ικανότητες να είναι αξιόπιστο συνομιλητή προ κάθε κατεύθυνση. σα ευχαριστώ. Το λόγο Κυρία Πρόεδρε, κυρία και η συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί τη νομική βάση για το διορισμό ειδικού εντεταλμένου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί προβλέπει ότι το Συμβούλιο δύναται με αίτημα τη ύπαρξη εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική να διορίσει ειδικό εντεταλμένο που θα αναλάβει εντολή για συγκεκριμένα θέματα πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την αρχή ήταν υπέρ τη αξιοποίηση αυτή τη ευκαιρία που δίνει η Ευρωπαϊκή Συνθήκη και πολλά και συζητήσαμε το διορισμό του ειδικού εντεταλμένου. Είχαμε και σχετικό ψήφισμα στα πλαίσια της ετήσιας έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο του 2009 και του 2010, καθώς και στην Ευρωπαϊκή, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής για το θέμα αυτό. Γι' αυτό και είμαστε ε, αναφανδών υπέρ της ε, σύσταση προς το Συμβούλιο για το διορισμό του ειδικού εντεταλμένου και τη έκθεση Αλαφράγκα. Και το λέμε αυτό με κάθε ειλικρίνη, γιατί αυτή ήταν η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σβένσον για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ θετική η απόφαση για το διορισμό του ειδικού εντεταλμένου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καλό θα ήταν επίσης να υπήρχε ε, μια παρόμοια θέση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένας παγκόσμιος, ας πούμε, εκπρόσωπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, θα πρέπει να προωθήσουμε επίσης ε, και θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη σταθερότητα σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να μιλήσουμε για τον εκδημοκρατισμό, Πρέπει να μιλήσουμε επίσης και για πολιτικά, πολυκομματικά συστήματα, αντί να μιλάμε μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο ειδικό εντεταλμένος θα έχει ένα καθήκον, μια αρμοδιότητα απίστευτα βαριά. Του ευχόμαστε, του εκπροσώπου αυτού, να καταφέρει να τροποποιήσει κάποιες ε, πραγματικότητες. Αν και δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο ο άνθρωπος αυτός να επιφέρει μια κάποια αλλαγή σε τεράστιες χώρες που έχουν τέτοια προβλήματα όπως η Κίνα ή η Ινδία. Επίσης, όταν μιλάμε για αυτά τα δικαιώματα, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο σεβασμός του ατόμου, ο σεβασμός της ακαιρεότητας του, του ατόμου. Τούτου λεχθέντος, εδώ εμείς στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η φήμη μας, βασίζεται, η μας βασίζεται και στην προώθηση αυτών των δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Ε, ο κ. Μίτσελ για 1,5 λεπτό ή 1 λεπτό. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Βαρόνια Άστον για την ευγένειά της και αυτής και του προσωπικού της και πολύ λυπάμαι που ορισμένοι ευρωβουλευτές ε, χρησιμοποιούν τα προνόμια τους για να σας μιλήσουμε αγένεια. Επίσης, διαφωνώ με τους συναδέλφους που εξέφρασαν την άποψη ότι ο ειδικό εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να είναι δικηγόρος. Το άτομο που θα διοριστεί, ούτως ή άλλως, θα πάρει ε, συμβουλές από δικηγόρους. Θα ήθελα ένα άτομο το οποίο να είναι αδέκαστο, θαραλέο, να έχει σωστή κρίση, να έχει ενέργεια και πάνω απ' όλα να μην ε, δεσμεύεται πολιτικά δεξιά ή αριστερά. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιέρετα. Δεν πρέπει απλώς να τα επιβεβαιώνει το δίκαιο. Θα πρέπει όλες οι πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθούν αυτό το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και ένα από τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η ισότητα ανδρών και γυναικών. Εκατό εκατομμύρια γυναικών λείπουν από αυτόν τον κόσμο. Γιατί, Γιατί ε, έγινε έκτρωση ε, των εμβρίων αυτών μόνο και μόνο επειδή ήταν ε, θηλυκά. Θέλω κάποιος να εμφανιστεί σε αυτό τον οίκο με θάρρος και να μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Για να μας μιλήσει με τρόπο θαραλέο, αδέκαστο και να μας πει ότι θα προωθήσει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα, γιατί είναι αδιέρετα και γιατί ε, δεν θα πρέπει καθόλου να, οι προκαταλήψεις να προωθούν κάποια και να γνώουν κάποια άλλα. Ευχαριστώ κυρία Νεντέλσεβα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Άστον, αγαπητέ συνάδελφοι. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Σαλαφράγκα διότι παρουσιάζει συνθετικά όλες τις ιδιότητες που πρέπει να καλύπτει η θέση αυτή. Πρόκειται για έναν από τους νομικούς στυλοβάτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή τα άρθρα 20. 21 και 23 και δεύτερον την εγγύηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, Ευρωπαϊκό, έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δράξει την ευκαιρία που του δίνεται επί ενός μέρους της νέας εξωτερικής πολιτικής της Ενώσεως και ελπίζω ο ρόλος του Κοινοβουλίου να ενισχυθεί και στη συνέχεια. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλούστατα για την θέση η οποία πρέπει να καλυφθεί από ένα δυναμικό άτομο αλλά το μήνυμα που θα δοθεί σε όλους τους περαιτέρω καταρχήν δηλαδή να προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία με ενισχυμένη εκπροσώπηση και με προώθηση αυτών των δικαιωμάτων διότι θα υλοποιείται στο νέο αυτό εκπρόσωπο και η κοινή μας πολιτική θα είναι πιο συνεκτική, θα προβληθεί περισσότερο, θα ενισχυθεί η προσπάθειά μας για ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν πρόκειται για μία απλώς τιμητική θέση, αλλά πρέπει να δοθεί μία ισχυρή εντολή για έναν πιο ελεύθερο κόσμο, όπου θα σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίδες. Ευχαριστώ. Το λόγο κύριο Γιακολίνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Άστον. Πράγματι αυτός ο ορισμός είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη, πιο αποτελεσματική, πιο χαρισματική, να φροντίσει και να ασχοληθεί με τους αδυνάμους, και η ύπαρξη ακριβώς αυτής της θέσης είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια και στον κύριο Σαλαφράνκα, τον πρόεδρο Σαλαφράνκα, για την ευθύνη που επέδειξε και το πνεύμα συνεργασίας. Έχουμε ανάγκη τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο τις δραστηριότητες αυτής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, και να δείξουμε θετικά βήματα προς τις τρίτες χώρες οι οποίες πολλά περιμένουν στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά για τις εμπορικές σχέσεις. Τώρα για τα θέματα της μετανάστευσης. Σήμερα τίθενται αρκετά θέματα τα οποία δεν έχουν λυθεί και που αφαιρούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτών οι οποίοι διαφεύγουν από καθεστώτα που καταπιέζουν τα δικαιώματά τους. Απέναντί τους θα πρέπει να επιδείξουμε σεβασμό. Τώρα για τα φυσικά δίκαια νομίζω ότι <clears throat> όλα αυτά συνδέονται με την προσωπικότητα του καθενός και γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει πλήρως τον ρόλο της και αυτός που θα επιλεγεί θα πρέπει δύο προϋποθέτης να πληρεί, να είναι μια προσωπικότητα θαραλέα και μια προσωπικότητα με χάρισμα. Ευχαριστώ η κυρία Κράτσα, ένα λεπτό. Η προάσπιση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, αποτελεί την βάση για την ε, εγκαθίδρυση αλλά και την λειτουργία της δημοκρατίας για την κοινωνική ειρήνη για την ανάπτυξη με συνοχή για τις ομαλές διεθνείς σχέσεις και γι' αυτό σωστά αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής της ένωσης. τα μέσα που διαθέτουμε ως τώρα ο πολιτικός διάλογος οι εμπορικές συμφωνίες με ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αποδειχθεί ότι δεν είναι επαρκείς γι' αυτό χαιρετίζω την πρωτοβουλία για τον ορισμό ειδικού απεσταλμένου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποστηρίζω τη σύσταση του κοινοβουλίου προς το συμβούλιο. νομίζω θα δώσει μια ορατότητα και συνεκτικότητα στην πολιτική μας. πρέπει ο ή απεσταλμένος ο ειδικός για τα ανθρώπινα δικαιώματα να μπορεί να κερδίσει την ανεξαρτησία της δράσης του αλλά και την ικανότητα ομαλής συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες με την κοινωνία των πολιτών με διεθνείς και περιφερειακές άλλες οργανώσεις. πρέπει παράλληλα να μπορεί να είναι ένας καλός ή καλή αναλυτής της πραγματικότητας στις διάφορες χώρες που δεν μας φτάνουν συχνά εμάς εδώ στο κοινοβούλιο οι πραγματικές συνθήκες. Ε, γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα γίνει μια σωστή επιλογή βλέπουμε τη σημασία που έχει και για τις καλές σχέσεις και την ειρήνη στον κόσμο η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα αραβικά κράτη που σε αυτή την πορεία του εκδημοκρατισμού υποφέρουν από τη μη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις διώξεις κατά των χριστιανών. πιστεύω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε μια συνεκτική και αποτελεσματική απάντηση και ο ορισμός του νέου αυτού θεσμικού προσώπου θα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Κράτσα. Περνάμε τώρα στη διαδικασία οφθαλμοθύρας και δίνω το λόγο στην κυρία Κορχολά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη. Υπήρξα μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στην χρονική στιγμή που ετέθη το θέμα αυτό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά νομίζω ότι εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά, μια πλειάδα προβλημάτων. Τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την Κίνα, παραδείγματο χάρη. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι λένε τι θα κάνει αυτός ο, ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα Είναι πάντα ένα θέμα το οποίο είναι, θεωρείται δευτερεύον. Όχι, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα να λαμβάνονται πάντα υπόψη με σοβαρό τρόπο και να είναι στο προσκήνιο. Κυρία Άστον, είπατε ότι η πρόθεσή σας είναι να βασίσετε όλες τις ενέργειές σας σε ένα επίπεδο συνεργασίας. Αυτό είναι σωστό. Δεν θα πρέπει να δούμε να υπάρχει, να υποσκάπτονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν υπήρξαν ποτέ τόσο σημαντικά ούτε προκάλεσαν τόσες αλλαγές και γεγονότα όσο τώρα. Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική δείχνουν τη σχέση μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατία. Επομένω, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αλλάξει την οτροπία τη σε σχέση με τι χώρε τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή για να μπορέσει να δει με ποιο τρόπο μπορεί να προωθήσει τη μετάβαση σε ένα δημοκρατικό καθεστώ και την οικοδόμηση εθνικών κρατών που να περιλαμβάνουν και το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι οι χώρες αυτές έχουν θυγεί από τα προηγούμενα καθεστώτα τους. Γι' αυτό το λόγο ο, η, η μελλοντική εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να είναι ένας σημαντικός συνομιλητής και των ΜΚΟ στις χώρες αυτές και των εθνοτικών μειονοτικών ομάδων θα πρέπει να μπορεί να κρατήσει επαφές με τα Ηνωμένα Έθνη και με τρίτες χώρες. Ο κύριος Όμπερ Μάιερ, για ένα λεπτό. Ούντερ Μάιερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι αρμοδιότητες του ειδικού αντιπροσώπου καλύπτουν πολλά θέματα. Είναι ευρύτατες αρμοδιότητες. Θα πρέπει να είναι περιορισμένος στα βασικά ε, προβλήματα. Μόνο για τα προβλήματα της Τουρκίας, η Σαρία, στη Συρία, συγγνώμη, η Σαρία, τα, οι ε, εκεί θα μπορούσε να ασχοληθεί ένας ε, ε, ειδικό αντιπρόσωπος ειδικά για αυτό το θέμα. Αν θέλουμε πραγματικά να καταφέρουμε κάτι, καλό είναι λοιπόν να επικεντρωθούμε στα βασικά. Δεν μπορεί να είμαστε πρωταθλητές σε όλα, γιατί θα χάσουμε. Ούτε θέλουμε να κατηγορηθούμε για ψεύδο δράσεις. Uh, report refers to freedom of expression, including on the internet. Η έκθεση αναφέρεται στην ελευθερία έκφρασης. Εδώ και λίγο καιρό ο Επίτροπος για Εσωτερικές Προθέσεις είχε ζητήσει να διωχθεί το συγκεκριμένο κόμμα λόγω ακριβώς του περιεχομένου της ιστοσελίδας του. Πολλοί φυλακίζονται γιατί δημοσιεύουν ερετικές απλά σκέψεις με ηλεκτρονικό τρόπο. Η ελευθερία έκφρασης είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως και η ελευθερία φυσικά του να μπορεί κανείς να διαβάζει και να ακούει το τι λένε οι άλλοι. Η Βρετανική κυβέρνηση προετοιμάζει ένα νόμο που δίνει τη δυνατότητα στις υπηρεσίες ασφαλείας να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται οσδήποτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν κάποιος από την κυβέρνηση σαν παράδειγμα μάθει ότι κάποιος σαν παράδειγμα επισκέπτεται ένα απαγορευμένο πολιτικό κόμμα τότε μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η θέση του στο δημόσιο. Και αυτό ισοδυναμεί και με αντίστοιχες ανελεύθερες ενέργειες για την απαγόρευση πολιτικών κομμάτων σε χώρες όπως το Βέλγιο. από μια χώρα όπου εκατοντάδες χιλιάδες ατόμων ζουν και εργάζονται σε κοσμικές συνθήκες. Ακόμα όμως αυτή η χώρα, η Ουγγαρία δεν είναι στον τρίτο κόσμο, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες μας δουλεύουν σε γραμμές ε, συναρμολόγησης για ξένες εταιρείε για περίπου 250 ευρώ το μήνα, σε αποθήκες, σε εργαστήρια, πάλι για 250 ευρώ την, το μήνα, μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη να απολυθούν, δεν έχουν καμία νομική προστασία <clears throat> σε ό,τι αφορά το εργασιακό δίκαιο. Το ερώτημά μου λοιπόν προς την κυρία Άστον είναι το εξής και θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρξει και μία εξαίρεση από τους κανόνες και να δώσει πραγματικά απαντήσεις στα αυτά αυτά. Ο νέος αυτός εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αντιμετωπίσει και περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι, θεωρείτε ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Οι μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λοιπόν στην Ουγγαρία θα εξεταστούν από τον ε, ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ποια διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μορβάη. Βεβαίω, κυρία Άστον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλα τα μέλη που συμμετείχαν στη συζήτηση ε, με τόσο ζήλο και ενθουσιασμό από όλες τις πολιτικές ομάδες για το θέμα αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας παραπέμπω στην έκθεση του κυρίου Σαλαφράγκα και στην εντολή του ειδικού ε, αντιπροσώπου και το δικό μου που είναι εξωτερική εντολή. Όπου είναι δυνατόν θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα και ε, γραπτός όσα δεν θα μπορέσω να απαντήσω τώρα. Γνωρίζω πολύ καλά ότι στη συζήτηση αυτή Πολλές ιδιότητες αναφέρθηκαν για αυτόν τον τόσο ενάρετο άνθρωπο που θα πρέπει να είναι ο ειδικό αντιπρόσωπος και συμφωνώ με πολλά από αυτά που ελέγχθησαν. Πράγματι αναζητούμε κάποιον δυναμικό, θαραλέο, πρόθυμο να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και να εκπροσωπήσει σωστά αυτόν τον ε, ρόλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά θέματα πρέπει να ε, δούμε με ευαισθησία, με πραγματική κατανόηση. Ε, βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να βρούμε 100% ε, προσαρμογή στην πραγματικότητα. Ε, θα πρέπει και στις πολιτικές δηλώσεις και οι πολιτικές δηλώσεις να ληφθούν υπόψη και οι συνθήκες. Είπαν πολλοί ότι είναι ο πρώτος θεματικός ειδικό αντιπρόσωπος και είναι σημαντικό να βρούμε τρόπους να εργαστεί σωστά. Αυτή θα είναι μια συνεχιζόμενη συζήτηση και είναι σημαντικό να μπορούμε να ε, ξανααναθεωρούμε ε, κάποια θέματα και να παντούμε στο Κοινοβούλιο. Σίγουρα θα οικοδομήσουμε στο έργο που ήδη υπάρχει και θέλω να αποτίσω φορό τιμή σε πολλούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις αντιπροσωπείες του που δουλεύουν πολλές φορές κάτω από δυσχερέστατες συνθήκες και ε, παρόλα αυτά κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να κάνουν το καλύτερο έργο. Και εν τέλει ο λόγο των συγητή μα, τον κύριο Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπάτη εκπρόσωπη τη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίε και κύριοι, θέλω να εκφράσω την ευαρέσκειά μου για το έργο που έχουν κάνει πολλοί συνάδελφοι για την προετοιμασία αυτή τη εργασία και είμαι ευγνώμων για όλε τι παρεμβάσει και τι συνεισφορέ αυτών που έλαβαν το λόγο σε αυτή τη συζήτηση. Με ικανοποίηση, κύριε Άστον, καταγράφω τη στεναρή σα δέσμευση ότι ο ειδικό εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μια συνεχή σύνδεση με αυτό το κοινοβούλιο σε σχέση με τους όρους εντολής που συζητήσαμε κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη δημοκρατική ρήτρα που έχουμε με τρίτες χώρες και ε, μου άρεσε πάρα πολύ η παρέμβαση του κυρίου Μίτσελ και όλα αυτά μου θυμίζουν την ιστοριούλα αυτή που αναφέρεται στον Αριστοτέλη πριν στον 4ο αιώνα όταν είχε τους ε, μαθητές του στην περιπατητική σχολή. Και όταν υπήρξε μια παρατήρηση η οποία δεν άρεσε στους φοιτητές του, ο Αριστοτέλης είπε δεν τα είπα εγώ αυτά, τα είπε ο Πλάτων, ο δάσκαλός μου. Αυτά λοιπόν είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται και στην τεχνολογική εποχή του ίντερνετ. Εγώ είμαι φίλος του Πλάτωνα, αλλά είμαι πιο πολύ φίλος της αλήθειας. Και επίσης και αυτό λοιπόν πρέπει να αντανακλάται και στην θεσμική δομή του εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει πάνω απ' όλα, πέρα από το να είναι φίλο του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να είναι φίλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι ώστε αυτές οι θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν στο 21ο αιώνα σε όλε τι περιοχέ του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. Πέρασε τη συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο στις 11 η ώρα. Στην μέση διάταξη έχουμε τώρα τη δήλωση της Αντιπροέδρου και υπά του εκπροσώπου για τα θέματα ασφάλειας και την εξωτερική πολιτική.